να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 16, παράγραφος 5. Υπέρ. Κατά. E eh, Απορρίπτεται. Τροπολογία 17, παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 παράγραφος 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 παράγραφος 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 20 στην ε, παράγραφο 14β υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 στην παράγραφο 15. Υπέρα Όχι. Λέει η Πρόεδρος. Το ψηφίζουμε. Ο συνάδελφος Ρουγκάης. Ευχαριστώ. να συζητήσει με τον συνάδελφο Μέγερ, έχουμε αλλάξει θέση για να διευκολύνουμε την ψήφιση της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 21, παράφος 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 στην παράγραφο 16. Η συνάδελφος Όκεν. Ε, δεν, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, ότι δεν συζητάμε τις τροπολογίες. Διότι συνειδητοποιώ ότι οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει πως το θέμα είναι πως είναι ωφέλιμο με μονομένα άτομα να συνυπογράψουν μια αναφορά γιατί μπορεί να ωφεληθούν όταν θίξουν μια μεγάλη υπόθεση ας πούμε εναντίον μιας μεγάλης εταιρείας ενώ μόνοι τους δεν μπορούν να σταθούν. Γι' αυτό και λέω πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερες συνεδριάσεις και να συζητήσουμε, να μπορούμε να συναντηθούμε. Ελπίζω να το υποστηρίξετε. Ψηφίσουμε για τροπολογία 22 παράγραφο 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Emendamento 23 al 17. Favorevoli. 23 στην παράγραφο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 στην παράγραφο 17α ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 παράγραφος 17α νέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 παράγραφος 18α νέα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 27, παράγραφος 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, παράγραφος 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 29, στην παράγραφο 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 30, στην παράγραφο 23. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 31 στην παράγραφο 23α νέα. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32, παράγραφος 23α νέα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33, ε, στη παράγραφος 23β, ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34, παράγραφος 24, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35, παράγραφος 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36, παράγραφος 24, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται, διορθώνει η Πρόεδρος. 37, στην παράγραφο 27, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 38, στην παράγραφο 27α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε να ελέγξουμε. Και ψηφίζουμε και πάλι στην τροπολογία 38, παράγραφος 27α, υπέρ. Ε, ε, Εγκρίνεται.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 11 11 eh, è respinto chi si astiene Αποχές. Vi, chiedo scusa. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή ήταν πριν ε, διαφορετικά τα νούμερα, ε, θεωρούσα δεδομένο ότι η 11 ήταν η πλειοψηφία. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 39 στην παράγραφο 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 στην παράγραφο 30α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 στην παράγραφο 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο του εγγράφου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται με δύο αποχές. means that Pascal has withdrawn her original in favour of this compromise. Possiamo passare all'esame degli emendamenti del progetto di relazione Bostinaro sulla biodiversità. Περνάμε τώρα στην εξέταση των τροπολογιών για την έκθεση Μποστινάρου για τη βιοπικιλότητα la votazione sugli emendamenti al documento. Emendamento 1 al paragrafo. Τροπολογία 1, παράγραφος 3α. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική, στην παράγραφο 5. Συνάδελφοι Μποστινάρου και Γκρούνη. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία, κυρία Πρόεδρε. Εγώ μαζί με τη συνάδελφο, την κυρία Γκρούνη, προτείνω να διαγράψουμε το τελευταίο τμήμα. Τη φράση που λέει δηλαδή το πιθανό αντίκτυπο σημαντικών έργων υποδομής που σχεδιάζεται στη Γαλλία για την κοιλάδα του Λίγυρα. Oui. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία με αυτή την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές. Ε, γκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η επόμενη και περνάμε άμεσα στην τροπολογία 3. Στην παράγραφο 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ripetiamo la votazione favorevoli contrari κατά respinto απορρίπτεται α όχι Δύο φάσεις. Favorevoli. Υπέρ, ξαναμετράμε. Please vote, Mr. Yard. Please do it. Eh, he changed. Ok. Ok, quindi approvato. Εγκρίνεται λοιπόν. Κατά. Astenuti. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. 4 10. Τροπολογία 4, παράγραφος 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, στην παράγραφο 12. Υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 5 στην παράγραφο 12. Υπέρ. Ε, κοντράρι. Κατά. Αστενούτη. Αποχές. Approvato. Emendamento 6 al παράγραφο 13. Favorevoli. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε επί του συνόλου του κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές, συνάδελφο Γκρούνη. Τελική ψηφοφορία για το έγραφο. Είστε υπέρ. Υπέρ. Ποιοι είναι. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται το κείμενο. Κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μποστινάρου. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και δεύτερον η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας και την ανάγκη να ενεργοποιηθεί η Ευρώπη και να προστατεύσει τη βιοπικιλότητά της. E Σας ευχαριστούμε και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το 19 την έκθεση σχετικά με τη διευρυντική επίσκεψη στην Ουέλβα. Υπάρχει έτοιμο να αναβληθεί η εξέταση αυτού του θέματος από πλευράς της κυρίας Γκρούνη. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να λείψω για λίγο στην Επιτροπή Απασχόλησης γιατί παρουσιάζω μια ανέκθεση εκεί και είναι τώρα τώρα. Οπότε θα ξαναέλθω μετά για να σας παρουσιάσω την Ουέλβα. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει να καθυστερήσουμε λίγο την εξέταση αυτού του θέματος και να πάμε στο 20 πρώτα. Η 1300 του 2007 που έχει υποβληθεί από τον κύριο Σίλα Μόρις. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Quindi do direttamente la parola per la Commissione ad Adam Nagy. Good Εκπρόσωπος της Επιτροπής. Καλημέρα σας από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Για αυτή την ε, αναφορά η Κομισιόν ήδη έχει κάνει ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι στα πλαίσια των, ε, της ΕΕΦΑ έγινε διαβούλευση για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Ο αναφέρον αποφάσισε λόγω του κόστους ότι δεν θα αλλάξει την απόφαση. Σε, δεν θα το προσπάθησε να το αλλάξει σε δικαστικό επίπεδο. Η Κομισιόν δεν αναφέρει κανένα, καμία πράξη η οποία να αποτελεί παράβαση. Και όπως ε, είπα, στην απάντηση του 2008 που έδωσε η Κομισιόν, ε, υπήρχε μια σε εξέλιξη υπόθεση εναντίον της Ιρλανδίας, μια δράση δηλαδή που ανελήφθη από την Κομισιόν δυνάμει του άρθρου 258 της συνθήκης. Η απόφαση του 10 βγήκε, αποστάλει, αποστάλει τον Ιούλιο του 2009 και μιλούσε για, την, για τις πολιτικές δράσεις και το κόστος. Για την, στο άρθρο 3.7 της ε, οδηγίας 35 αναφέρονται οι διατάξεις για το κόστος αυτών των διαδικασιών, το οποίο δεν πρέπει να είναι απαγορευτικά υψηλό. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των απαγορευτικά, αυτού του απαγορευτικού υψηλού κόστους ε, αναφέρεται και στο κομμάτι που λέει ότι... Συγγνώμη, συγγνώμη. Ζητώ κυρίες και κύριοι να είσαστε στη θέση σας για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι και άλλοι παρακαλώ να καθίσετε και να είσαστε στις θέσεις σας. Ε, Συνεχίστε παρακαλώ. Το δικαστήριο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της αρχής ο Ριπένο πληρώνει στο Ιρλανδικό σύστημα, στο Ιρλανδικό νομικό σύστημα και είπε ότι τα Ιρλανδικά δικαστήρια μπορούν να αρνηθούν σε ένα, ατυχές, σε ένα αποτυχόν μέλος να, ε, να ε, αναλάβει το κόστος και αυτό είναι διακριτική η μεταχείριση από το δικαστήριο. Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, σωστή εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σχετικό άρθρο. Και εκτός αυτού, στη συνέχεια η Κομισιόν άρχισε συζητήσεις με τις Ιρλανδικές Αρχές ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι ε, κανόνες αυτοί ή θα ενσωματωθούν στο ελλανδικό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάποιος θέλει να παρέμβει. Αν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, τότε από ό,τι βλέπω κλείνει εδώ αυτή η αναφορά. Και περνάμε στο σημείο 21 τώρα. Αναφορά 353-2009 Λουίτζι Ντε Μαρίνο Ιταλικής υπηκότητας Ο κύριος Πάκερ θα λάβει τον λόγο Thank you and good morning. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους σας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη απάντησε γραπτός σε αυτή την αναφορά αυτό που θα θέλαμε εδώ να πούμε και να κάνουμε είναι να τονίσουμε ότι στο έγγραφο το οποίο είχε σταλεί στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Αναφορών στη 2η Μαρτίου 2009, ότι αυτό το έγγραφο πράγματι <clears throat> είχε αφορούς την ε, ε, υπηρεσία περιβαλλοντικών μελετών στην καμπάνια στην Ιταλία και στάλει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερωτικά. Δεν είχε στραφεί σαφώς προς το Κοινοβούλιο αλλά μόνο παράπλευρα. Το έγγραφο αφορά την απουσία δημόσιας διαβούλευσης για μια μελέτη ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον στο Καστέλ Βολτούρνο, σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία του 2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει ότι θα ενημερώνονται οι πολίτες για τις ε, δράσεις ε, των μελετών αυτών, των εξεταστικών αυτών ενεργειών. Δεν αναφέρεται όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους πολίτες και έτσι το σημαντικό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι η μεταφορά από τις Ιταλικές αρχές αυτής της πρόβλεψης έχει ξεπεράσει εκείνα τα πλαίσια τα οποία προβλεπόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ζήτησε ο αναφέρον να ξαναρχίσει, να ξανανοίξει η διαδικασία μελετών για το περιβάλλον και των επιπτώσεών τους και σε σχέση με την ακύρωση της προηγούμενης ε, αυτής ε, με την με την Alta Tutela στα Ιταλικά. Όμως ε, δεν έχει νομική βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτό το θέμα, διότι το θέμα καλύπτεται από εθνική νομική διάταξη. Γι' αυτό αν υπάρχει κάποια παράβαση ή παραβίαση, είναι θέμα εθνικής μεταφοράς στο δίκαιο αυτό από την Ιταλία και όχι θέμα παραβίασης ευρωπαϊκού δικαίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κάποιος θα ήθελε να παρέμβει παρακαλώ. Αν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, θεωρείται ότι κλείνει και αυτή η αναφορά. Σημείο 22, αναφορά 128-2009 του Νόμπερτ Κάιζερ. Έχει τον λόγο η κυρία Πέτρα Σότ, παρακαλώ. Θα αναβάλουμε λοιπόν, μια και δεν ε, υπάρχει αυτή η παρουσία. Περνάμε στο θέμα αναφοράς 23. Ε, εντάξει. Υπάρχουν προβλήματα με όσους θα έπρεπε να είναι παρόντες. Θα προτείνουμε μια διακοπή 10 λεπτών για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά από 10 λεπτά συνεδρίασή μας. Συμφωνείτε, εντάξει. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται και πάλι η συνεδρίασή μας. Παρακαλώ καθίστε. Eh, λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση όσον αφορά το σημείο 22. <clears throat> Αναφορά <clears throat> τη που έχει υποβληθεί. Δίνουμε τον λόγο στην κυρία Σότ. Κυρία Πέτρα Σότ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση πρώτα απ' όλα. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη σαφήνεια να εκθέσω τα θέματα. Ο Κάιζερ παραπονείται για το ότι στη Γερμανία στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών της ε, ε, Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας και των κρατηδίων οι επιδοτήσεις ε, για τα οικογενειακά επιδόματα δεν καταβάλλονται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει γάμος αλλά όπου υπάρχει καταχωρημένη συμβίωση εταίρων όπου με τον ίδιο τρόπο έχει ρυθμιστεί το θέμα σε σχέση με τη Γερμανία όπως στην Λέει ότι είναι θέμα ίσης μεταχείρισης. Το να μην αντιμετωπίζεται ισότιμα η συμβίωση με το γάμο είναι παραβίαση της οδηγίας που προστατεύει από, μη, από την μη δικαιολογημένη αρνητική διακριτική μεταχείριση. Υπάρχει λοιπόν έτοιμα εδώ να υπάρχει ισότιμη αναγνώριση ε, συμβίωσης και επίσημου γάμου. Το 10 ε, τοποθετήθηκε σε μια γερμανική περίπτωση όπου επρόκειτο για την, ε, το επίδομα ε, χειρίας και αναφερόταν ότι έτοιμα ισότιμης αντιπα... αντιμετώπισης υπάρχει μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο γάμος σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση επιδόματος δηλαδή χειρίας είναι θέμα εθνικών δικαστηρίων να διαπιστώσουν το τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημείο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία παραβάση κατά της Γερμανίας για τη μη πλήρη υλοποίηση της αντίστοιχης οδηγίας ξεκίνησε αυτή η διαδικασία το 2007 και αυτό το σημείο εξακολουθεί να μένει ανοιχτό. Αυτό το σημείο πρέπει δηλαδή η καταχωρημένη σχέση συμβίωσης στην, στα ιατρικά επιδόματα, στην ε, ε, σύνταξη χειρίας και στα οικογενειακά επιδόματα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται και βρισκόμαστε στην περίοδο, στην συγκυρία τώρα του να δούμε αν θα καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 10 ασκώντας προσφυγή αυτό εκκρεμεί. Νομικά δεν είναι απόλυτα σαφή τα πράγματα, επειδή όπως προανέφερα αυτό το θέμα, αν πραγματικά σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα ο γάμος και η καταχωρημένη σχέση συμβίωσης με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, επειδή είναι ταυτόσιμα θέματα, είναι ακαθόδες θέμα. Το ΔΕΚ δεν το αποφάσισε, το άφησε στα κράτη-μέλη, στα δικαστήρια των κρατών μελών να αποφασίζουν. Γι' αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομικά δεν είναι απόλυτα σαφές το πώς μπορεί μπορεί να ληφθεί μια απόφαση. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις γερμανικές αρχές. Μια απόφαση εφέτος θα πρέπει να ληφθεί, θα ληφθεί. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι υπάρχει ένα σχέδιο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας για μια τροποποίηση, μια αλλαγή σε αυτό το σημείο. Αν γινόταν πραγματικότητα αυτό το νομοθέτημα, τότε σε ομοσπονδιακό επίπεδο τα προβλήματα τα οποία αναφέρει ο κύριος Κάιζερ θα επιλειόντουσαν. Δεν ξέρω όμως αν τα ομοσπονδιακά κρατήρια θα ακολουθούσαν μια τέτοια κατεύθυνση. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο η περίπτωσή του θα είχε επιληθεί. Όμως υποθέτω ότι και τα κρατήδια κατά κανόνα αντίστοιχα θα ρυθμίσουν αυτά τα θέματα ώστε η δική του περίπτωση μ, πιθανότατα μελλοντικά θα επιληθεί. Όχι όμω αναδρομικά. Από κάποιο χρονικό σημείο θα παίρνει αυτό το οικογενειακό επίδομα. Αυτά είχα να πω. Ε, ευχαριστούμε πολύ. άλλε παρεμβάσει, παρακαλώ εσεί. Η πρότασή μου θα ήταν γι' αυτό, επειδή ο διάλογος προφανώς μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους μέλους στη Γερμανία δεν έχει ολοκληρωθεί, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι ότου να έχουμε κάποια περαιτέρω στοιχεία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε επαφή και να δούμε πότε ο διάλογος αυτός θα ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, μέχρι ολοκλήρωση του διαλόγου, να παραμείνει ανοιχτή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη παρέμβαση. Bien, yo estoy de acuerdo. Εντάξει, συμφωνώντας με αυτή την παρέμβαση μετά και από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά στη συνέχεια και γι' αυτό περνάμε στη συνέχεια τώρα Εντάξει, περνάμε λοιπόν στο σημείο 23 τώρα. Αναφορά 363-2008 Ντόρις Μούλερ. Θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος της Επίτροπης ο κύριος Μάρτιν Γκάστερ παρακαλώ. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή η περίπτωση αφορά πιθανή αρνητική διακριτική μεταχείριση αλλοδαπών όσον αφορά φόρο ε, για ακίνητα σε σχέση με την Ελλάδα. Η κυρία Μούλερ, η αναφέρουσα που ζούσε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και που είναι Γερμανίδα υπήκος, αποφάσισε να αγοράσει από κοινού με το σύζυγό της ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Υπό κανονικέ συνθήκες θα εξαιρεί από το 11% μεταφοράς ε, αγοράς ε, ιδιοκτησίας ε, ως φόρου διότι ήταν μόνιμα κάτοικος της Ελλάδας πράγμα το οποίο είναι η προϋπόθεση που επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο όμως, σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι ελληνικές αρχές απέτυσαν την υλοποίηση και μιας άλλης προϋπόθεσης, ενός άλλου όρου, για να μπορεί να τύχει αυτής της εξαίρεσης από τον φόρο. Και αυτός ο όρος ήταν ότι έπρεπε να είχε εργαστεί στην Ελλάδα επί ένα έτος πριν από την αγορά αυτού του ακινήτου, του εν λόγω ακινήτου. Τώρα, αν αξιολογήσουμε νομικά αυτή την προϋπόθεση, αυτόν τον όρο, πρέπει να ομολογήσουμε πράγματι ότι αυτός ο όρος αποτελεί μια παραβίαση ε, ευρωπαϊκού νόμου, ευρωπαϊκής νομικής διάταξης. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας πλήρως αναλύσει τα στοιχεία της ελληνικής νομοθεσίας 1078 ε, όσον αφορά την ε, φορολογία ε, αγορών ακινήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η απέτηση δεν απορρέει από το ίδιο, τον, ίδιο αυτόν νόμο και ούτε εμπεριέχεται σε αυτόν νόμο και έτσι δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει ότι υφίσταται γενική διοικητική τέτοια προσέγγιση και έτσι λοιπόν με βάση αυτό θα μπορούσε να ασκηθεί κάποια ε, προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώς δεν μπορεί σε σχέση με τέτοια θέματα να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, διότι δεν υφίστανται νομικά τα μέσα με τα οποία θα μπορούσε να παρέμβει και να αναμειχθεί στις ε, εσωτερικές νομικές και διοικητικές διαδικασίες. Και έτσι, για αυτούς τους λόγους οι διατάξεις που αφορούν την εθνική νομοθεσία πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει την αναφέρουσα σε μια επιστολή Δεκεμβρίου 2008 σχετικά. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι αυτός ο νόμος 1078 του 1980 είχε αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, βάση μια, ένα άλλο παράπονο, μια άλλη καταγγελία. Άσκησε ε, την προσφυγή επί παραβάση κατά της Ελλάδας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση στοιχεία τα οποία άμεσα εμπεριέχονται σε αυτόν τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση κιόλας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ και τον Μάιο εφέτος 2010 είχαμε την πρώτη ακροματική διαδικασία στο ΔΕΚ για αυτό το θέμα. Αυτή η περίπτωση του 10 αφορά όπως προαναφέρθηκε άλλες νομικές διατάξεις Πρώτον, την απέτηση να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ζητήθηκε η εξαίρεση αυτή σε σχέση με την Ελλάδα να μπορεί να ισχύει και για αγοραστές που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν εκεί. Και η δεύτερη πτυχή σχετικά είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα χορήγησε αυτή την εξαίρεση σε Έλληνες υπηκόους Παρότι όμως ε, η απέτηση μόνιμης εγκατάστασης δεν υλοποιείται σε σχέση με αυτούς. Όσον αφορά όμως ε, την αναφέρουσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να ζητήσει να δοθεί συνέχεια σε αυτή την υπόθεση στα εθνικά δικαστήρια της Ελλάδας. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ευχαριστώ κάποιος που θέλει να παρέμβει. Εσείς παρακαλώ. Τίθεται το ερώτημα εδώ. Γνωρίζουμε αν η αναφέρουσα αυτή την νομική δυνατότητα την έχει χρησιμοποιήσει τη σύσταση δηλαδή σε σχέση με το, την επιστολή του 2008 που συστάθηκε η διαδικασία να συνεχιστεί σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικά δικαστήρια. Έχουμε πληροφορία αν το έκανε αυτό ή όχι, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή την υπόθεση, αυτή την αναφορά. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να τύχει συνέχεια στα εθνικά δικαστήρια και από αυτή να απορρέουν τα ε, περαιτέρω συμπεράσματα μετά. Λοιπόν, το θέμα Γνωρίζουμε αν έκανε η αναφέρουσα κάτι σχετικά στα εθνικά δικαστήρια της Ελλάδας και θα μπορούσαμε λοιπόν μετά να πούμε ότι κλείνουμε αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας ενημερώσει την αναφέρουσα δεν είχε κάποια άλλη επαφή. Δεν γνωρίζουμε αν ακολούθησε αυτή τη νομική οδό η αναφέρουσα ή όχι. Äh, äh, και επίσης ε, η αναφέρουσα δεν μας έχει γνωστοποιήσει αν επιτυχώς, αν στέφτηκε με επιτυχία το εγχείρημά της ή όχι. Πρόεδρος. Πιστεύω κυρίε και κύριοι ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να απευθύνουμε μια επιστολή στις ελληνικές αρχές <clears throat> σε σχέση με αυτό το θέμα. Απλά και μόνο μια επιστολή της Επιτροπής Αναφορών προς τις ε, ελληνικές αρχές ε, εκφράζοντας το ενδιαφέρον μας. Να δούμε πώς βλέπουν επίσης πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα οι ελληνικές αρχές. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου. Συμφωνείτε με αυτήν. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 24 στη συνέχεια. Αναφορά 242-2007 Lars Evan Γιόργενσεν. Θα λάβει τον λόγο Michael Μεντούνα, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Thank ah, ευχαριστώ. Η αναφορά έρχεται από την Δανία, από έναν Δανό υπηκό, ο οποίο είναι παντρεμένο με μια Βραζιλιάνα και αποφάσισε να θέλουν να ζήσουν στην Σουηδία. Αναφέρει λοιπόν ότι η σύζυγό του θα πρέπει να λάβει άδεια εργασία για να μπορέσει να εργαστεί στην Δανία. Τονίζω ότι το ζευγάρι μένει μόνοι νόμιμα στην Σουηδία. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν δικαίωμα να κινούνται και να εγκαθίστανται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ε, ζευγάρι αυτό εξασκεί αυτό το δικαίωμα αυτή τη στιγμή, διαμένοντα στη Σουηδία. όλα αυτά, μια, επειδή ο υπήκος μένει στην Σουηδία, όλα τα δικαιώματα εγκατάστασης αφορούν το σουηδικό δίκαιο ως προς αυτό. Η νομολογία του δικαστηρίου πρόσφατα, το Μάρτιο 2006, C-05, ΜΑΤΕΝ και C Cottage, λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η υπήκος του τρίτη, της τρίτης χώρας έχει δυνατότητα να εργαστεί χωρίς ε, προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς να ε, χρειάζεται άδεια εργασία. Μόνο στο κράτος μέλος το οποίο ζει και εργάζεται, δηλαδή τη Σουηδία. Επομένως, η σύζυγος από τη Βραζιλία έχει κάθε δικαίωμα και δικαίωμα πρόσβαση στην ε, αγορά εργασία στην Σουηδία, αλλά οι Δανέζικε αρχέ σωστά είπαν ότι αν αυτή θέλει να μετακομίσει στη Δανία και πρέπει να εργαστεί στη Δανία, θα πρέπει να έχει ε, άδεια εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Όκεν. Ε, ε, κοίταξα αυτή την περίπτωση, αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν διαφωνώ με την δανέζικη νομοθεσία και είναι πολύ περιοριστική όσον αφορά την... Δεν μπορώ να παραβώ την δανέζικη νομοθεσία εδώ. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ως απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αδύνατο για μένα να πω ότι αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει στη καλύτερη σύνταξη νομοθεσίας. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρος, θεωρούμε λοιπόν ότι κλείνει αυτή η αναφορά. Σωστό. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Και περνάμε τώρα στην αναφορά 25. Συγγνώμη. Στην ημερήσια διάταξη το 25, 448 αναφορά 2008. Από τα αρχικά έχουμε εδώ ΚΑΑ Πολωνικής Ιθαγένειας αναφέρον. Ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής που παρενέβη προηγούμενα, κύριος Μεδούνα, παρακαλώ. Thank ε, πάλι σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αφορά προβλήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση αιτήσεων υπηκών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γαλλία. Ε, ισχυρίζεται ο αναφέρον ότι οι γαλλικές αρχές πήραν πέντε μήνες για να εκδώσουν ένα τέτοιο πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα το στοιχείο του Ευρωπαϊκού ε, Νόμου σε αυτή την περίπτωση είναι η Οδηγία σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, οικείων τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία έπρεπε να μεταφέρει αυτή την οδηγία μέχρι τον Απρίλιο 2006. Το έκανε αυτό η Γαλλία και πράγματι το άρθρο 8 της οδηγίας απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δίνουν τέτοια πιστοποιητικά εγγραφής επιτόπου άμεσα να μπορούν να τα εκδίδουν. Και όσα, όπως αναφέρει αναφέρουσα, δεν συνέβη αυτό όσον αφορά τη δική της ατομική περίπτωση. Εξετάσαμε, ελέγξαμε σε σχέση με τα θέματα της γαλλικής νομοθεσίας τα σχετικά και βρήκαμε ότι Πράγματι η ε, γαλλική νομοθεσία σωστά μετέθεσε και μετέφερε αυτές τις διατάξεις της οδηγίας και καταρχήν όλες, η, ε, όλα τα πιστοποιητικά αυτής της εγγραφής ε, χορηγούνται στην Γαλλία άμεσα αυτό ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση λοιπόν μη ορθής εφαρμογής από τις γαλλικές αρχές όχι μόνο ευρωπαϊκού νόμου αλλά και εθνικού νόμου της Γαλλίας, της εθνικής νομοθεσίας και δεδομένου ότι το πιστοποιητικό αυτό εντωμεταξύ είχε εκδοθεί προς την αναφέρουσα και δεδομένου ότι ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση αυτή η καταγγελία, δεν έχουμε αντίστοιχα παράπονα, οι καταγγελίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να ανοίξει οποιασδήποτε διαδικασίες επί ε, προσφυγή κατά της Γαλλίας. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η γαλλική νομοθεσία βαίνει καλώς και ε, σωστά εφαρμόζεται. Ήταν μόνο μια ξεχωριστή, μονομένη περίπτωση αυτή. Εν τω μεταξύ έχει το πιστοποιητικό αυτό εκδοθεί και εν πάση περιπτώσει και η οδηγία και το ε, εθνικό νομοθέτημα στη Γαλλία διασφαλίζουν ότι ακόμα και χωρί ε, αυτέ ε, αυτά τα πιστοποιητικά έχουν δικαίωμα εγκατάσταση οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γαλλία άσχετα από το θέμα εγγραφή ή όχι. Δεν μπορούν να υπάρξουν λοιπόν αρνητικέ επιπτώσει για τα δικαιώματα της αναφέρουσας. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Εσείς ζητήσατε τον λόγο, παρακαλώ. Με βάση τα προηγούμενα που ακούσαμε, θα πρότεινα, μια στιγμή, θα πρότεινα να κλείσουμε αυτή την αναφορά, θα έλεγα. Θα πρότεινα λοιπόν να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Ε, πρόεδρος, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και εγώ ως Πρόεδρος θεωρώ ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κλείνει αυτή η αναφορά εδώ. Σημείο 26. Αναφορά 1039-2007 του Τζουζέπε Λιπάρη αναφέροντος. Θα λάβει τον λόγο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο κύριος Λαβρέντσος παρακαλώ. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα του νούμερου κλάουζους που διέπει την είσοδο στη τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου στην Ιταλία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, η, αρχικά η Επιτροπή σας είχε ε, θεωρήσει μη αποδεκτή αυτή την αναφορά γιατί το άρθρο 141 της συνθήκης που έγινε 162 με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας λέει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ισένωσης. Όμως οι αναφέροντες με, επανήλθαν με μια νέα επιστολή το Μάιο του 2009 με την οποία μάλλον, στην οποία προσάρτησαν ε, μία σύσταση από τις Ιταλικές Αρχές Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Αγοράς και εκεί αναφέρεται μία σύσταση όπου αναφέρεται ότι ο αριθμός των εισακτέων στις εν λόγω σχολές θα πρέπει να αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτή την σύσταση της αρχής του ανταγωνισμού. Επιθυμεί όντως η πρόσβαση ή η η στα πανεπιστήμια να είναι όσο γίνεται ευρύτερη. Φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στο επάγγελμα το ιατρικό και το διατρικό και από την άλλη πλευρά την παιδεία που θεωρείται δικαίωμα όλων και είναι ευρύτερη. Η Κομισιόν όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε δεν έχει νομικά δεσμευτικά μέσα για να κάνει οτιδήποτε άλλο αλλά επαναλαμβάνω, επιθυμεί ότι η πρόσβαση θα να είναι όσο γίνεται ευρύτερη και ότι η η παιδεία να διατίθεται σε όσο γίνεται περισσότερους ε, υποψηφίους και εφόσον δεν έχουμε νομικό μέσο για να ενεργήσουμε θα οδηγηθείτε μάλλον να κλείσετε αυτή την ε, αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. ¿Alguna intervención? Κάποιοι που θέλουν να παρέμβουν παρακαλώ. Λοιπόν, θεωρούμε ότι κλείνει και αυτή εδώ η αναφορά επίσης. Βλέπουμε από το Προεδρείο, ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την έκθεση της κυρίας Γκρίνη για την Βουέλβα. Κάποιος όμως απουσιάζει από την Επιτροπή ο κ. Μποστινάρου που ήταν στην επίσημη αντιπροσωπεία. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι σε σχέση με τους αναφέροντες και σε σχέση με τις παρούσες αρχές θα έπρεπε να υπάρχει κάποια δράση από πλευρά μας θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Γκρίνη για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα αυτού του πρώτου εγγράφου για την επίσκεψη που είχαμε κάνει εκεί ε, στην Βέλβα Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σα ζητήσω να με συγχωρήσετε γιατί χρειάστηκε να πάω στην Επιτροπή ε, Απασχόληση ε, ζητώ συγγνώμη λοιπόν που σας ανάγκασα να αλλάξετε κάπως την ημερήσια διάταξη. Όντως λοιπόν τον Φεβρουάριο πήγαμε στην Βέλβα και πριν είχαμε επίσης σταματήσει στη Σεβίλη με συνόδευση σε αυτή την ε, ε, αποστολή η κυρία Όκιν και ο κύριος Βοστινάρο και βεβαίως ο κύριος Μέγερς από τους μη επισήμους. Ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους ε, του Υπουργείου Βιομηχανία και Περιβάλλοντος, με ε, του ετού αναφέροντε. Έπειτα τη δεύτερη μέρα πήγαμε στην Ουέλβα ε, και είδαμε και επισκεφθήκαμε την εταιρεία που έχει δεχθεί τα πύρα και καθώς και του συνδέσμους για την προστασία του υγείας. Ε, συναντηθήκαμε τελευταία μέρα με τον δήμαρχο του Έλβα, και εκπροσώπους της περιφέρειας της Ανδαλουσίας. Είδαμε λοιπόν πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα ρήπανσης στον χώρο αυτό. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα ΜΜΕ. Το θέμα, η αντιπροσωπεία μας, η αποστολή μας ε, τα πήγε πολύ καλά. Η υποδοχή ήταν ικανοποιητικότατη από τις διάφορες αρχές με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή. Αλλά αλήθεια που είναι ένα ότι είναι ένα θέμα διόλου εύκολο. Για μας που δεν είμαστε επιστήμονες φυσικά, το, η δυσκολία είναι να έχουμε ταυτόχρονα μελέτες, να ακούσουμε και τους ε, ενδιαφερόμενους ε, για το θέμα, που έχουν απόψεις ε, κάποιες φορές ιδιαίτερα αποκλίνουσες. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε συστάσεις, καταλήξαμε σε συστάσεις βεβαίως, ελπίζουμε ότι θα μας ακούσουν και το πρώτο που διαπιστώσαμε ήταν ε, μια έλλειψη επικοινωνίας πραγματική ανάμεσα σε όλες τις αρχές ε, εθνικές, ε, δημοτικές, περιφερειακές και πιστεύω πως όλοι θα πρέπει να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι καθώς και οι αναφέροντες ε, και η εταιρεία, αλλά και οι τοπικέ σύνδεσμοι για την προστασία της υγείας με ειδικού που θα μπορέσουν πραγματικά να είναι αρκετά αντικειμενικοί και να απαντήσουν στα όσα ε, τους ρωτούν, αλλά και που να είναι και συμπεφωνημένοι από όλους. Δηλαδή, μόνιμος διάλογος θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί για να κατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνη και να καθησυχαστεί και ο πληθυσμός. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ε, στην ε, περιοχή αυτή, ωστόσο ο πολίτης δεν γνωρίζει σίγουρα τα όσα έχουν γίνει. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί και το θέμα της προηγούμενης ρήπανσης που κατά την άποψή μου ο χώρος θα πρέπει να καθαριστεί, να εξεταστούν τα προβλήματα του ποταμού και από σήμερα να προσέχθει ώστε η εταιρεία να ακολουθήσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες που είναι κοινοτικέ οδηγίες. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει η εταιρεία αυτή ε, επιπλέον να απαντήσει στα αιτήματα των αναφερόντων, διότι πιστεύω και εμείς το ζήσαμε ότι δηλαδή η επιχείρηση δεν είχε δώσει την έγκρισή της για να επισκεφθούμε με τους αναφέροντες ε, το χώρου της. Ε, αυτό το σεβαστήκαμε αφού δεν είχαμε την έγκριση, ήταν λογικό, αλλά πιστεύω πως η διαφάνεια είναι πάντοτε καλύτερη και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν μπορούν να ε, εκτεθούν και προς τους άλλους. Φυσικά η ρήπανση είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται δεχτό και υπάρχουν τώρα μέσα για να εργαστούμε με σεβασμό στο περιβάλλον μεγαλύτερο. Πιστεύω πως αυτή η έλλειψη λοιπόν διαφάνειας και η έλλειψη επικοινωνίας είναι βάση για το πρόβλημα. Θα συστήνουμε επίσης να γίνουν μελέτες, αλλά με οργανισμούς που να είναι απόλυτα αντικειμενικοί και να μπορούν να είναι αποδεκτοί από όλες τις πλευρές. Ε, συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν μελέτες για το έδαφος και για το νερό. Και νομίζω επίσης πως ε, σε αυτό το χώρο υπάρχουν ε, πολλές, παλαιές αποθηκεύσεις φωσφογύψου Για... Θα πρέπει να καθαριστεί λοιπόν το έδαφος. Ε, θα υπάρχουν επίσης ε, ε, κομματερές οικιακών αποβλήτων που δίνουν ιδιαίτερα άσχημη όψη στον χώρο και που δίνουν και άλλη εικόνα γιατί όταν κανείς δεν γνωρίζει τη βιομηχανία φωσφογύψου φτάνει σε μια επιτερία, σε μια επιχείρηση, σε ένα χώρο που εξαιρετικά βρώμικο πράγμα το οποίο δίνει κακή εικόνα και φοβίζει, τρομάζει σίγουρα και πιστεύω πως η επιχείρηση αλλά και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε ο χώρος να καθαριστεί. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την αρχή του παίρνουν πληρώνει. Άρα αυτό θα πρέπει να το δούμε με την εταιρεία, με την επιχείρηση. Εγώ υποστηρίζω τη βιομηχανία γιατί είναι θέσει απασχόληση. Ήρθαμε σε επαφή, συναντηθήκαμε με του υπαλλήλου και με τα συνδικάτα που φοβούνται για το κλείσιμο του εργοστασίου ε, και ειλικρινά για κάθε πολιτικό είναι δραματικό το να χρειαστεί να κλείσει ένα εργοστάσιο. Αντίθετα, μπορούμε να ζητήσουμε από την επιχείρηση να σεβαστεί το περιβάλλον. Γιατί αυτό που πρέπει να ε, δούμε είναι ότι αν κλείσει η επιχείρηση θα πάει αλλού η παραγωγή. Θα πάει αλλού, στον πλανήτη μας πάλι, ίσως και να είναι και εκτός ένωσης, Δηλαδή, ίσω αυτό να μα ικανοποιεί και να πούμε να εμεί ησυχάσαμε. Εγώ προσωπικά, όταν σκέφτομαι το περιβάλλον, δεν σκέφτομαι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά την υδρόγειο. Δηλαδή δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει μια τέτοια, τέτοιου είδους λύση που απλώς θα μετακινηθεί η ρήπανση αλλού. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπέρ λοιπόν του κλεισίματο. αντίθετα να είμαστε υπέρ τη αρχή ορυπαίνων πληρώνει, να γίνουν έλεγχοι τυχαίοι και απροειδοποίητοι στις εταιρείε. στη Γαλλία το κάνουμε αυτό πολύ, για να ελέγξουμε αν όντως σέβονται το σύνολο των οδηγιών και των νόμων που ισχύουν. Και καλό τι αρχέ, ε, τις εθνικές, τις περιφερειακές, τις τοπικές να κάνουν τέτοιους προειδοποίητους ελέγχους. Εάν τυχόν χρειαστεί να κλείσει η εταιρεία αυτή, θα πρέπει να επιβληθεί σε αυτήν να συμμετέχει στην αποκατάσταση του χώρου. Να δούμε πώς μπορεί να δημιουργηθούν εκ νέου θέσεις απασχόλησης με σεβασμό στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά. Ε, νομίζω πως έχω αναφέρει τα πάντα εδώ και είμαι στη διάθεση όλων και ελπίζω πως οι συνάδελφοι θα συμβάλλουν επίσης. Ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ το σύνολο των Ισπανικών Αρχών και του συναδέλφου της Αντιπροσωπείας. Και φυσικά να ευχαριστήσω και το προσωπικό που μας συνόδεψε από τη Γραμματεία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κρίνη για αυτή την εκτενή παρουσίαση, περιεκτική παρουσίαση και τώρα θα είναι πολύ χρήσιμη σε σχέση με αυτή την παρουσίαση και το έγγραφο. Θα έχουμε χρόνο να ξεκινήσουμε συζήτηση και να υπάρξουν παρεμβάσεις ε, για να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Παρούσα είναι η κυρία Γκερέρο, πρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας του Δήμου της ε, Γουέλβα. Καλώς ήρθατε εξ ονόματος Επιτροπής Αναφορών. Και στη συνέχεια θα έχουμε την σχολίαση και θα λάβουν τον λόγο και οι αναφέροντες και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι θα αρχίσει ο γύρος των παρεμβάσεων στη συνέχεια από πλευρά ημών Ευρωβουλευτών. Η κυρία Γκερέρο έχει τον λόγο λοιπόν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για τον Δήμο της Βουέλβα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συνεδρίαση που θα συνεισφέρει χωρίς αμφιβολία να ρίξει άπλετο φως για ένα θέμα που πάντα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη προσοχή λόγω της, ε, των κοινωνικών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν και των επιπτώσεων που φυσικά στη δική μας ε, περιοχή όλα όσα αφορούν την ε, μόλυνση και τη ρήπανση είναι πολύ σημαντικά. Και καθώς προερχόμαστε από τη Γουέλβα, όπως είπα, είναι σημαντικό να μπορούμε να είμαστε παρόντες σε αυτή τη συζήτηση. Χωρίς αμφιβολία, πολύ σημαντική η συζήτηση για ένα θέμα που εκπροσωπούμε εμείς στο Δήμο μας ε, εδώ σήμερα. Η καταγγελία, η αναφορά που μας έχει συναθρήσει εδώ μπορεί να είχε νόημα πριν από 20-25 χρόνια κύριε και κύριοι. Σήμερα όμως δεν έχει νόημα αυτή η κατηγορία, η ε, καταγγελία ή αναφορά μπορεί να έχει κάποιες ε, σκοπιμότητες που εξυπηρετεί και εξηγούμε η περιβαλλοντική πραγματικότητα της Βέλβα δεν έχει καμιά σχέση σήμερα σε σχέση με πριν από 20-25 χρόνια δεν έχει καμιά σχέση μεταξύ άλλων λόγω της βούλησης των επιχειρήσεων και των ε, διοικήσεων και των αρχών και των πολιτών της Βουέλβα. Ε, Μια βούληση στεναρή και μόνιμη να κάνουμε διαφορετικά πια τα πράγματα σε σχέση με το όπως γινόντουσαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Και μπορούμε να ε, θέσουμε σε 20 χρόνια στο παρελθόν το σημείο καμπής. Από το σημείο εκείνο οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις επομίστηκαν την αρχή της προσέγγισης της αηφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης αυτή την αρχή θέλω να τονίσω και να αναβαθμίσω την αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή νοοτροπίας να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου της Βουέλβα. Αληθεύει ότι εδώ και 20 χρόνια κυρίες και κύριοι ξεκινούσαμε από μια κατάσταση που ήταν σαφές ότι μπορούσε να βελτιωθεί και ήταν και ανησυχητική κιόλα πρόεδρε. Όμως επίσης αληθεύει ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη την πραγματικότητα πριν από 20 χρόνια. Υπήρξε σημαντική αλλαγή στην υφή των πραγμάτων πραγμάτων. Πράγμα το οποίο κάνει άδικο σήμερα να εντοπίζεται στην Ιουέλβα ως μια ιδιαίτερα μολυσμένη περιοχή. Και είναι άδικο αυτό, επειδή λίγες περιοχές υπάρχουν στην Ευρώπη που να έκαναν τέτοια τεράστια προσπάθεια. Τόσο ειλικρινή και αποφασιστική προσπάθεια για να ενταχθεί η νοοτροπία και ο πολιτισμός της αηφόρου ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στις παραγωγικές διαδικασίες. Και έτσι να μπορέσει η ανάπτυξη να ευθυγραμμίζεται με τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Κυρίε και κύριοι, ακριβώ ε, στον 21ο αιώνα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι προσπάθειε που έγιναν τι τελευταίε δεκαετίε. Προσπάθειε που έδωσαν τη δυνατότητα να είναι ορόσημο σήμερα η Γουέλβα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου όμω να κάνω εδώ μια διακοπή για να σα δώσω κάποια στοιχεία που θα σα βοηθήσουν να καταλάβετε την πραγματικότητα στην επαρχία μα, στην περιφέρειά μα. Κυρίε και κύριοι, πάνω από ένα τρίτο τη περιοχή τη Γουέλβα προστατεύεται με τον ένα ή άλλο τρόπο νομικά. Στην Γουέλβα έχουμε 23 φυσικού χώρου που προστατεύονται. Από αυτού ένα εθνικό πάρκο, δύο φυσικά πάρκα και οκτώ δρυμούς ε, φυσικούς προστατευόμενους δρυμούς. Έχουμε το εθνικό ε, πάρκο του Ντονιάνα που είναι κληρονομία τη ανθρωπότητα τη UNESCO και έχουμε και το ε, φυσικό πάρκο τη Σιέρα Ντε και των κορυφών Αρότσε και κυρίες και κύριοι θα έλεγα ότι αυτά τα οποία σας περιέγραψα δεν πιστεύω ότι είναι η πραγματικότητα πραγματικότητα μιας περιοχής ιδιαίτερα μολυσμένης. Και έτσι πρέπει ακριβώς να δούμε ότι υπάρχει μια ειδική πραγματικότητα σήμερα που είναι ε, ο σεβασμός του περιβάλλοντος. Όπως προανέφερα, έκανε τεράστια προσπάθεια η Γουέλβα για να ενταχθεί στον πολιτισμό της αηφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κύριες δραστηριότητες οικονομικές της επαρχίας μας είναι ο τουρισμός, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η γεωργία και όλοι έχουν εστερνιστεί την βιώσιμη ανάπτυξη και την αηφορία. Μια και είναι περιορισμένο ο χρόνο σε πέντε λεπτά για την παρέμβασή μου και θέλω να σεβαστώ αυτό το όριο, θα αναφερθώ μόνο Στι βιομηχανικέ δραστηριότητες, στην προσπάθεια που έγινε για να εξυγχρονιστούν οι παραγωγικές διαδικασίες και για να πετύχουμε μια οικονομική δραστηριότητα που θα σέβεται το περιβάλλον το φυσικό περιβάλλον. Οι χημικές βιομηχανίες της ε, επαρχίας μας ε, κατά τη διάρκεια 1993-2008 500 ε, εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν για να προσαρμοστούν οι παραγωγικές διαδικασίες στο σεβασμό του περιβάλλοντος. 500 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το στένος της βούλησης και την αποφασιστικότητα των βιομηχανιών να σεβαστούν το περιβάλλον. Περισσότερες μελέτες, περισσότερε, αν θέλετε πιο εμβαθυμένα στοιχεία που μπορούν να συλλεγούν, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι έγιναν όλα αυτά. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και όλα κατέδειξαν ότι η κατάσταση όσον αφορά τη μόλυνση, τη ρήπανση τη επαρχία τη Γουέλβα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πιο αυστηρές αναλύσεις. Έγιναν μελέτες από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, από το Πανεπιστήμιο της ε, Γουέλβα, από την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Όλες αυτές οι έρευνες είχαν θετική έκβαση. Μέχρι ποιο σημείο θα γίνεται αυτό. Ποια έκθεση πρέπει να είναι ικανοποιητική για να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων. Είναι αυτονόητο ότι από πλευρά των διοικήσεων, ιδιαίτερα τη κυβέρνηση τη Ανδαλουσία, συμμετείχαν στη συνεισφορά και στη χρηματοδότηση αυτών των βελτιώσεων ακολούθησαν τις βιομηχανίες. Πάρα πολλά πράγματα τα συνόδευσαν όσον αφορά την βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας της Γουέλβα και υιοθέτησαν δεσμεύσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ανυποχώρητη βούληση να είμαστε όσον αφορά το περιβάλλον, να σεβόμαστε το περιβάλλον. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποια προσωρινά προβλήματα, βρίσκονται, αν θέλετε, στην επίλυσή του. Πρόκειται να επιληθούν. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει παναχώρηση, δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Βρισκόμαστε στην ορθή κατεύθυνση και έτσι, χωρί καμία διακοπή, άοκνα εργαζόμαστε για να εξυγχρονιστούν οι παραγωγικέ διαδικασίε και να υπάρξει βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Και έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την καταγγελία αυτή τη αναφορά. Ιδιαίτερα όσο αφορά την ε, ε, κοινωνική επίπτωση που έχουν τέτοιου είδου στοιχεία. Θα ήθελα να πω κυρίε και κύριοι ότι αυτή η καταγγελία και αυτή η στάση μπορεί να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε στρατηγική. Σε μια στρατηγική όμω που δεν έχει καμιά σχέση με το να υπάρξει δικαιοσύνη για την επαρχία τη ε, Γουέλβα. Μπορεί να προκαλέσει κοινωνικέ ε, ταραχέ ή συναγερμό. Όμω εμεί θεωρούμε ότι μια ε, δημοτική αρχή όπω η δημοτική αρχή τη Γουέλβα δεν θα πρέπει να θεωρήσει με κανένα τρόπο δίκαια αυτή την κατάσταση αντιμετώπιση της δικής μας περιφέρειας. Στη Γουέλβα κάναμε καλή δουλειά πιστεύω. Κάναμε σωστά τη δουλειά μα και τα καθήκοντά μα. Και έτσι είμαστε βέβαιοι ότι οπωσδήποτε μπορούν να βρεθούν κάποια θέματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Είναι όμω πρόσκαιρα και προσωρινά αυτά τα προβλήματα και μπορούν να βρουν τη λύση του. Και έτσι έχει προβλεφθεί μια λύση για όσα θέματα εκκρεμούν. Είναι σαφέ λοιπόν κυρίε και κύριοι και γνωρίζουμε προ τα που πορεύονται τα πράγματα στο μέλλον. Και έχουμε προπαρασκευαστεί ώστε να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Και ολοκληρώνω. <clears throat> Θέλουμε να το κάνω, θέλω να το κάνω όπω ξεκίνησα την παρέμβασή μου με αφορμή σε σχέση την, την μετάβαση της ε, Επιτροπής Αναφορών στη Γουέλβα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για μια σοβαρή δουλειά που έγινε, μια μέθοδο εργασίας που δίνει μια εγγύηση για μας, εγγύηση ότι η τελική έκταση αυτού του οργάνου είμαι πισμένη ότι θα είναι πολύ προσεκτική και πάρα πολύ ε, αντικειμενική. Μια έκθεση που θα δίνει δίκαιο στις προσπάθειες που έγιναν από την διοίκηση του Δήμου της Βουέλβα προσπάθειες που έγιναν κατά τις τελευταίες ε, δεκαετίες για να προσαρμόσουμε τις παραγωγικές διαδικασίες στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσει. Απαιτήσεις νομοθετικές αλλά και για τους πολίτες μας. Προσπάθεια που έδωσε την ευκαιρία να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, βιομηχανικής ανάπτυξης και του σεβασμού στο περιβάλλον. Υπόδειγμα, πρότυπο αυτό και έτσι για την αηφορία και τη βιώσιμη οικονομία του μέλλοντος. Βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Μπορεί κάποια πράγματα να πρέπει να βελτιωθούν. Εντάξει. Όμως όχι περισσότερο από τις χώρες που είναι γύρω μας και τους γείτονές μας. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε και πώς να κάνουμε τα πράγματα. Και θα το κάνουμε με ε, αίσθημα υπευθυνότητα και ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για αυτήν την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να δώσουμε τον λόγο στους αναφέροντε που μπορούν να παρέμβουν. Πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα παρεμβαίνω εκ νέου σε σχέση με την πλατφόρμα ε, της ε, Γουέλβα από πλευράς αναφερόντων και μάλιστα με εντολή 25.000 ατόμων που ενέκριναν πολύ πρόσφατα <clears throat> όχι πριν από δεκαετίες εντάξει, αλλά πολύ πρόσφατα ενέκριναν και προσυπέγραψαν την αναφορά μας. Το κάνω αυτό πρώτα απ' όλα για να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη ατομικά εξ ονόματός μου και το κάναμε ήδη γραπτός προς την κυρία Γκρούνη για το συμβάν εκείνο το οποίο έγινε όσον αφορά την επίσκεψή σας. Να ξέρετε ότι στη Γουέλβα πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν μαθαίνοντας ότι δεν επετράπει η επίσκεψη στην ε, ε, βιομηχανία αυτή όσον αφορά την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορούσαν να βλέπανε από πρώτο χέρι με κάθε διαφάνεια αυτά που οι αναφέροντες ε, ήθελαν να σας θέσουν υπόψη και ήταν θα μπορούσε να είναι αποσαφινιστικό και θα μπορούσε να γίνει αυτή η επίσκεψη με συνοδεία των εκπροσώπων της βιομηχανίας για να δείτε εκεί τα απόβλητα <clears throat> και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό σε σχέση με εκείνου που κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όχι επί δεκαετίε, αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών δώσαμε ολόκληρο αγώνα για να, σταματήσουν, να σταματήσει αυτή η μόλυνση, η ρήπανση αυτή. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η, τα απόβλητα του ε, ε, φωσφογύψου ε, θα τερματιστούν σύντομα. Αυτό αποφασίστηκε από μια απόφαση εθνικών δικαστικών αρχών που καθορίζουν την 31η Δεκεμβρίου 2010 ως τελική ημερομηνία προθεσμία. Πάνω από πέντε χρόνια λοιπόν ήταν εκείνα. Τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια, όχι δεκαετίες όπως αναφέρθηκε εντάξει, τα τελευταία πέντε χρόνια μιας νομικής ε, διαδικασίας όπου η Φερτιβέρια έχανε κάθε ένα και όλους τους πόρους που είχε ασκήσει δικαστικά κατά της εντολής της Γενικής Αρχής Προστασίας των Ακτών, της Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος που είχαν δηλώσει ότι έπαβε να ισχύει η δυνατότητα άδειας ε, κατάθεσης αυτών των αποβλήτων στο περιβάλλον και που έτσι έπαβαν να ισχύουν τα όσα είχαν δοθεί με αυτή την άδεια. Κυρίες και κύριοι, χρόνια χρειάστηκαν, κύριοι Ευρωβουλευτές, χρόνια αγωνιζόμαστε τα τελευταία αυτά χρόνια που αγωνιζόμαστε απέναντι σε μια οικονομική εξουσία που είναι η Ένωση Χημικών ε, Βιομηχανιών της Γουέλβα. Απέναντι στην πολιτική εξουσία επίσης δώσαμε αγώνες και με την κυβέρνηση της ε, Ανδαλουσίας ε, και με το μέγιστο σεβασμό και με την εκπρόσωπο της κυρίας Προέδρου του Δήμου της Γουέλβα. Αγώνες δώσαμε και σε σχέση με την μεδιατική αυτή των, στα μέσα ενημέρωσης ε, ε, όσα συνεπάγονται έχουμε επίσης ε, αναφερθεί και έχουμε δώσει αγώνες. Ήταν χρόνια αγώνων αυτά, όπου οι πολίτες της Γουέλβα, 25.000 υπογραφές που ε, είχαν συναθριστεί για αυτή την αναφορά το Δεκέμβριο 2008 όχι πριν από δεκαετίες το Δεκέμβριο του 2008 αυτό δείχνει ότι έπρεπε να δώσουμε αγώνα εναντίον εκείνων που αγνοούσαν την πραγματικότητα 1200 εκτάρια των δημόσιων αυτών εκτάσεων ε, που από μια επιχείρηση ε, λιπασμάτων είχαν μολυνθεί από φωσφογύψο 120 εκατομμύρια ε, ε, κιλά από αυτό το υλικό και σε λίγα μέτρα απόσταση από την πόλη της Βουέλβα, Αυτή είναι η πραγματικότητα. 7.000 τόνοι των ε, τεφρών που έχουν μολυνθεί από το Κέσιο 237 που τοποθετήθηκαν σε αυτή την ελογενή περιοχή σαν να ήταν μια χωματερή και που κυρίες και κύριοι αυτό είναι μια πραγματικότητα στάχτες τέφρες ε, ε, σιλικίου ε, με υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού με καρκινογενή υλικά και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία αυτά κυρίες και κύριοι είναι σήμερα αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα υλικό το οποίο από το Πάλος de la Frontera είχε τοποθετηθεί εκεί, από την χημική βιομηχανία που ξεφορτώθηκαν σε αυτή την ελογενή περιοχή και μεταφέρθηκαν εκεί αντί να έχουν πάει στην ε, χωματερή αλλού. Αυτά είναι η πραγματικότητα των τελευταίων ετών στη Γουέλβα κάθε είδους στερεά απόβλητα, αστικά στερεά απόβλητα, που επί χρόνια από τον Δήμο της Γουέλβα απαιτήθεντο εκεί, είναι και ήταν στο παρελθόν μια πραγματικότητα για μας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, καταλαμβάνουν ένα εύρος, μια έκταση, όσο εκείνη που καταλαμβάνει η πόλη ίδια της Γουέλβα. Μια πόλη 148.000 πολιτών. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν σήμερα στην πόλη της Γουέλβα. Όχι της επαρχίας της Γουέλβα, της πόλης της Γουέλβα. Εντάξει. Χρόνια λοιπόν ολόκληρα που ανεχόμαστε αυτή τη μόλυνση που συνεχιζότανε. Πάσης φύσεως ρήπανση και μόλυνση. Μια κατάσταση που θέτει τη Γουέλβα σύμφωνα με μελέτες που έγιναν πολύ πρόσφατα υγειονομικά και όσον αφορά την υγεία όπως το Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάβρα στην Βαρκελόνη ή και το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης το θέτουν επικεφαλής, θέτουν την πόλη μας όσον αφορά τις περιπτώσεις ε, ε, καρκινογένεσης, ε, καρκίνη, αναπνευστικές ασθένειες και καρδιαγγειακές ασθένειες επιπλέον. Δεν, ε, ε, είμαστε εμεί οι οποίοι επινοήσαμε μια τέτοια πραγματικότητα. Δυστυχώ κυρίε και κύριοι αυτή είναι η ίδια η πραγματικότητα. Και η κοινωνική διάσταση και συνειδητοποίηση και όλες οι σφιγμομετρήσεις και μελέτες που δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους μήνες παρόλη την κατάσταση οικονομικής κρίσης που διατρέχουμε τοποθετούν το περιβαλλοντικό πρόβλημα ως το κυριότερο πρόβλημα το οποίο ανησυχεί τους πολίτες της Βουέλβα σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι προσδοκίες πολλών ατόμων της Βουέλβα που αγωνίστηκαν επί χρόνια και που συνεχίζουν να αγωνίζονται βρίσκονται στους ώμους σας. Έχουν αναποτεθεί σε εσά Πολλά βλέμματα έχουν στραφεί σήμερα εδώ στην Ευρωβουλή. Εγώ εξ ονόματος της πλατφόρμας της Ria de Huelva και των 25.000 ατόμων που προσυπέγραψαν το αίτημα της αναφοράς που καταχωρήθηκε το Δεκέμβριο 2008 σας ευχαριστούμε ειλικρινέστατα σας ευχαριστούμε για την απάντηση που δώσατε εσείς οι ίδιοι. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι οι προσδοκίες που έχουμε στο δικό σας όργανο και στα άτομα που επισκέφθηκαν από εσάς στη Γουέλβα ικανοποιήθηκαν και με το παραπάνω. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε με τις καλύτερες εγγυήσεις στο μέλλον θα είναι ο σεβασμός από πλευράς των Ισπανών, Ισπανικών αρχών, περιφερειακών αρχών και τοπικών αρχών της Ισπανίας και της Γουέλβα, σεβασμός της έκθεσης με όλα τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Θα είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει χρηματοδότηση που θα προέρχεται από όλες τις διοικήσεις και θα είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί όπως αναφέρεται στο ίδιο το έγγραφο να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων ώστε να μην επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Η κυβέρνηση της Περιφερειακής Αρχής της Ανδαλουσίας πρέπει να διασφαλίσει αυτή τη συμμετοχή της σήμερα σε όλα όσα συσχετίζονται με το θέμα της αποκατάστασης της μπάλσα της, του φράγματος των φωσφογυψικών υλικών και όπως και σε τόσες περιοχές της ε, Ευρώπης που υφίστανται τις επιπτώσεις ρήπανσης και μόλυνσης δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα ηθικής, ηθικό ζήτημα. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα από έναν ποιητή, τον Χουάν ε, ότι όσον αφορά μόνο εκείνους που νοιάζονται για τις αδρές γραμμές της οικονομίας υπάρχουν άλλοι που τους νοιάζει η λεπτή γραμμή της ζωής που πρέπει να είναι σεβαστή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή θεωρώ ότι η δράση της Επιτροπής Αναφορών για αυτό το θέμα καταδεικνύει την αξία της Επιτροπής Αναφορών. Ήταν μια επιτυχία αυτό. Κατέδειξε ότι ο ρόλος των αναφερόντων μπορεί να επικεντρώνεται σε ένα θέμα και μπορεί η δική μας Επιτροπή να είναι διαμεσολαβητής και τα αποτελέσματα είναι εξόφθαλμα και προφανή για όλους τώρα. Τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδωσαν δίκαιο στους αναφέροντες και τα δικαστήρια στην Ισπανία, όπως και το ανώτατο δικαστήριο, έδωσε εντολή να σταματήσουν οι εναποθέσεις αποβλήτων μέχρι τα τέλη του 2010 εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε και ανταποκρίθηκε με υποδειγματικό τρόπο και in situ επιτόπου και στην ε, διερεύνηση των γεγονότων. Και υπήρξε και τεκμηριωμένη έτσι γνωμοδότηση. Είμαστε λοιπόν σε θέση να μπορέσουμε να προσφύγουμε στο 10 για αυτό το θέμα. Πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί αναδιαδήποτε στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε και θέσπισε ότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας με αυτά τα απόβλητα δεν είναι ένα υποπροϊόν βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Όχι, είναι βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει να τύχουν μια σαφέστατης αποκάθαρσης μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε δεν αποκαθάρθηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό επειδή παραβιάζει την ε, οδηγία ΙΠΠΣ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτά τα απόβλητα ευρωπαϊκά, ε, βιομηχανικά με συγχωρείτε, επικίνδυνα απόβλητα που συσσωρεύονται δίπλα στην πόλη της Βουέλβα... είναι πιθανόν να υπήρχαν περιπτώσεις πιο επικίνδυνες ακόμα αποβλήτων σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια όμως ο κίνδυνος αυξάνεται με τη σόρευση. αυξάνονται οι κίνδυνοι όσον αφορά το περιβάλλον και το σώμα μας. Είναι αυτά απόβλητα και υπολείμματα επικίνδυνα βιομηχανικά όπως και τα όσα βρίσκονται γύρω από το Εθνικό Πάρκε του Ντονιάνα. Είναι μια περίπτωση όπου υπήρξε χωρίς οποιαδήποτε αντίδραση που πολλούν οι αρχές ε, τα, ε, φωσ... φωσφογυψή σαν να είναι κάποιο ε, παράγωγο βιομηχανικών δραστηριών, δραστηριοτήτων. Βρήκαν όμως από πλευράς της Guardia Civil οι υψηλότατες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που μολύνουν και τις σοδιές όσον αφορά τους γεωργούς κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Ντονιάνα. Αυτό δεν είναι επινόηση ή εφεύρημα λοιπόν, αλλά πραγματικότητα. Κυρία εκπρόσωπε του Δήμου της ε, ε, Γουέλβα, μπορεί κανείς να, ε, να μπορέσει να πλύνει το πρόσωπό του, όχι, δεν μπορεί όμως να ξεπλύνει τα απόβλητα αυτά. Δεν είναι θέμα εξοραϊσμού ή αισθητική. Άλλο θέμα είναι τα βαρέα μέταλλα, τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Και αυτό το οποίο πιστεύουμε και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, δεν είναι δυνατόν να γίνει απλόν ένα ξέπλυμα αυτών των αποβλήτων. Έχουμε εκατοντάδες εκτάρια φωσφογύψων που, έχουν, φωσφογύψων που έχουν σήμερα μολύνει το περιβάλλον. Δεν είναι το να υπάρξει ε, κάποια δυνατότητα να ε, υπάρξει κάποια, κάποιο χορτολίβαδο που θα φυτρώσει πάνω από αυτές τις ε, ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων και έτσι όλα θα ξεχαστούν Πρέπει να μην υπάρξουν τέτοιε ε, ε, αποθέσεις ε, αποβλήτων, να μην, υπάρξουν, να μην υπάρξει η μόλυνση του ποταμού της Γουέλβα και όταν αναφέρονται τα στοιχεία για τα πάρκα ή τα στοιχεία προστατευόμενων περιοχών γύρω από τη Γουέλβα έχουμε και το ίδιο το θέμα της προστασίας της Βουέλβα, Όποιος μολύνει πληρώνει. Σε περίοδο οικονομικής κρίση από πλευρά τη Ισπανία δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνει η επιχείρηση αυτό το οποίο πληρώνουν όλοι οι Ισπανοί πολίτες και όλοι οι Ευρωπαίοι. Πρέπει λοιπόν οι υπεύθυνοι να κληθούν να πληρώσουν. Απευθύνουμε έκκληση και ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με τη διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ενθαρρύνουμε να υπάρξουν ανεξάρτητες μελέτες, μελέτες διότι σε σχέση με τις μελέτες όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ίδιων των εργαζομένων την ε, Τιβέρια με τα ίδια μέσα έγιναν της βιομηχανικής αυτής εκμετάλλευσης ή ε, με κάποιους οι οποίοι είχαν ε, σχέση άμεση με αυτή την επιχείρηση. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους μελέτες. Χρειάζονται ανεξάρτητες μελέτες, αντικειμενικές ανεξάρτητες μελέτες, ώστε να έχουμε και την δυνατότητα να παρέμβουν και αλλοδαπά ε, ερευνητικά ιδρύματα όπως της Γαλλίας που βρήκαν υψηλότατες ε, συγκεντρώσεις ε, επικινδύνων δηλητηριωδών στοιχείων στην Γουέλβα. Αυτό πρέπει να γίνει όσον αφορά την προστασία και του περιβάλλοντος και των πολιτών της Γουέλβα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές, έχουμε εμπιστοσύνη στην δράση των πολιτών που οδήγησε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έδωσε ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα πώς πρέπει κανείς να δρά και να ανοίγει τις θύρες των θεσμικών οργάνων για να μπει μέσα το φως να φωτιστεί το θέμα της υγείας των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε ίσως την Κομισιόν τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά θέτει δύο πτυχές, δύο σα, επί των οποίων υπήρξε διεξοδική πληροφόρηση προηγούμενα. Αφενός αφορά την πιθανή κακή εφαρμογή της οδηγίας 96, 1996 Ευρατών όσον αφορά την υλοποίηση των κυριότερων στοιχείων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την προστασία των πολιτών όσον αφορά βλαπτικές ουσίες. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο επεξηγήθηκε επαρκώς με προηγούμενες δράσεις ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση και με τις, ε, τα όσα θα έπρεπε να εκπονηθούν σε μεγαλύτερο βάθος. Όμως η αναφορά επιπλέον έχει και μια άλλη συνιστόσα που είναι η συνιστόσα της κακής εφαρμογής και εκτέλεσης της οδηγίας για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το σημείο στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια έρευνα που οδήγησε σε μια ταυτοποίηση παραβίασης ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας τριών οδηγιών αφενός της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, δεύτερον της οδηγίας IPPS και της ε, οδηγίας όσον αφορά τις ε, χωματερές και τις, ε, και τις ουσίες. Και για αυτές τις τρεις όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, εκείνο το οποίο ερευνάται είναι συγκεκριμένα και χειροπιαστά η εναπόθεση αυτών των ε, προϊόντων φωσφογύψου στην ελογενή περιοχή ε, της Γουέλβα ώστε να μην μπορεί αυτή η χωματερή να δημιουργήσει πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Όμω, υπό το πλαίσιο αυτή τη οδηγία εξετάζεται το αν οι αρμόδιε αρχέ λαμβάνουν ή έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν ώστε τα απόβλητα εκεί τα οποία συσσωρεύονται θα μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα δημόσιο ε, όργανο που θα διαχειρίζεται αυτά τα ε, απόβλητα και θα μπορεί έτσι να τα ελέγξει. Αυτό όσον αφορά την, το χώρο απόθεσης, εναπόθεσης. Υπάρχει και μια νέα έρευνα η οποία αφορά την εφαρμογή της οδηγίας IPPC και η οποία έρευνα στοχεύει στο να διαπιστώσει αν η λειτουργία, όχι η εναπόθεση, η λειτουργία αυτή τη φορά και η δράση των επιχειρήσεων που δρούν εκεί υλοποιούν, δηλαδή της Φερτιμπέρια και της FMC υλοποιούν τις διατάξεις εκείνες που έχουν υιοθετηθεί και υλοποιούν όλα τα προληπτικά μέτρα ελέγχου και πρόληψης όσον αφορά τις ε, ε συντεταγμένες διατάξεις. Εδώ κάνουμε λόγο για πηγάδα, πηγάδια, για εμπόδια, φραγμούς, ε, φράγματα τα οποία θα μπορούν να οδηγήσουν στο να προλάβουμε μια πιθανή ρήπανση ή μόλυνση. Και έτσι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξετάζεται αν συνάδουν με τις διατάξεις που υφίστανται και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τρίτον, έρευνα για το αν η οδηγία για τα απόβλητα υλοποιείται ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσει που έχουν μέχρι σήμερα διατυπωθεί. Όπως επισημάνθηκε η έρευνα ξεκίνησε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδοποιήθηκε σε σχέση με την πρώτη ε, φάση με μια ειδοποιητήρια επιστολή και λαμβάνοντας υπόψη την εξέταση των ε, ε, ε, ισχυρισμών αυτών από την, από την Ισπανική κυβέρνηση, τις Ισπανικές αρχές, ειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση ότι υπάρχει δυνατότητα άσκησης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εξετάσουμε είναι αυτονόητο με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία και τη έκθεση και τα συμπεράσματα τα οποία υποβάλλονται από την έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι λογικό ότι θα ενημερώσουμε την Επιτροπή Επιτροπή των Αναφερόντων για τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει και ο Wolfgang Kill από την Κομισιόν. Και έτσι ολοκληρώνεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής. Χωρίς μικρόφωνο. Uh, um. Ξέχασα να πω ότι έχουμε εδώ και την εκπροσώπηση μέσα Ρία de Huelva. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ αξιολογική έκθεση την οποία λάβαμε χτε. Ο συνάδελφο από την ε, ε, του Κομισιόν που ανέφεραν τα θέματα της ε, ακτινοβολίας από πέρσι. Ε, καλώς το έπραξαν. Ε, εμείς θα σας κρατούμε ενημέρωση, συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα και σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία θα τα προσθέσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ. Δίνω τότε το λόγο στον συνάδελφο Μέγερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκρίνη για την έκθεσή της. Πιστεύω ότι είναι μια έκθεση πάρα πολύ αντικειμενική σε σχέση με την περιγραφή της επίσκεψης και τις συστάσεις που αντανακλούν πλήρως θα έλεγα, θεωρώ εγώ, τα προβλήματα και πώς πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα αυτά σήμερα όπως έχουν. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας έκθεσης λοιπόν που είναι αυτονόητο ότι μπορεί να βελτιωθεί, όλα μπορούν να βελτιωθούν, αλλά που βαίνει προς την ορθή κατεύθυνση, στοχεύει στη σωστή κατεύθυνση. Οι συστάσεις αφορούν κάθε ένα και όλα τα στοιχεία όπου η κοινωνία των πολιτών και οι ίδιες οι αρχές της ε, Ισπανικής κυβέρνησης, το υπογραμμίζω αυτό, του Ισπανικού κράτους, οι αναφέροντες, ε, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιες οι αρχές θα πρέπει να επιλύσουν. Τι να γίνει λοιπόν με αυτά τα χίλια τόσα εκτάρια εκτάσεις που αυτή τη στιγμή είναι μολυσμένα. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή είναι η συζήτηση και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Χάρη στου ε, αναφέροντες, διότι οι αναφέροντες είναι εκείνοι που κατάφεραν αυτό το σημαντικό γεγονός. Σίγουρα στράφηκαν στην γραμματεία της Επιτροπής μια και υπάρχουν δύο συσσωρευόμενες ε, και που έχουμε τη Μέσα Ντελαρία. Λείπει όμως η πλατφόρμα της ΡΙΑ και αυτό η προσθήκη της, του ονόματος αυτό είναι και αυτό σημαντικό. Χάρη σε αυτούς τους αναφέροντες είπα, διότι αυτοί κατάφεραν ή βοήθησαν ώστε να δουλέψουμε προς την ορθή κατεύθυνση. Ποια προβλήματα υπήρχαν πρώτα απ' όλα αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε ή όχι να την, ε, κατάσταση με τα φωσφογύψη. Έλεγαν οι αναφέροντες όχι, δεν έπρεπε να συνεχίσουν να είναι αποτίθενται εκεί. Τα δικαστήρια του έδωσαν δίκιο και υπάρχει και η καταληκτική ημερομηνία. Δεκέμβριο 2010 λίγη καταλήγει η δυνατότητα αποθήκευσης φωσφογύψου. <clears throat> Αναφέρθηκε ότι δεν είναι υποπροϊόν βιομηχανικό τα φωσφογυψοειδή. Είναι ένα προϊόν όχι υποπροϊόν, είναι απόβλητο τοξικό βιομηχανικό και ως τοξικό απόβλητο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι υποπροϊόν ή υποαπόβλητο τοξικό. Είναι ένα απόβλητο τοξικό που πρέπει έτσι να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έδωσε δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες λέει δεν κάνουμε λόγο για υποπροϊόν αλλά για ένα τοξικό απόβλητο. Ως τοξικά απόβλητα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα φωσφογύψη. Αλλά επίσης οι αναφέροντες ζητούσαν από τις ε, ε, κυβερνήσεις και από τις τοπικές αρχές ε, όταν θα πάψουν να υπάρχουν τέτοιου είδους αποθέσεις αποβλήτων, ποια συνέχεια θα πρέπει να δοθεί. Και εδώ το Υπουργείο στην Ισπανία, το αρμόδιο Ισπανικό Υπουργείο, ήταν κατά και μας το είπαν αυτό και στην επίσκεψη κιόλας σε σχέση με την Φερτιβέρικα. Ήταν μια λύση, ας το πω έτσι, καλεσθητική εξοραϊσμού του περιβάλλοντος. Κάποια ε, δεντράκια να ε, μπορέσουν να φυτευτούν, κάτι να γίνει για την έκθεση. Ε, το αντίστοιχο Υπουργείο Περιβάλλον, για, Ισπανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασία των Ακτών είπε ήταν εναντίον. Προηγούμενα είπε πρέπει να υπάρξει υδρογεολογική χημική μελέτη, χημιολογική μελέτη, ραδιολογική μελέτη για να δούμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Και όταν θα γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά, τότε να ληφθεί δράση. Δεν είναι μικρή υπόθεση αυτή. Υπάρχει μεγάλη έκθεση και βαρέων μετάλλων και μόλυνσης ε, και για αυτούς τους λόγους λοιπόν οι αναφέροντες και το ίδιο το Υπουργείο συνέπεσαν στη συζήτηση σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκε σε αυτά η κυρία Γκρίνι και στα συμπεράσματα ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των αρχών. Συντονισμός μεταξύ των κρατικών αρχών, των τοπικών αρχών, περιφερειακών αρχών, μεταξύ όλων, ώστε με αυτά τα στοιχεία τα επιστημονικά, επιστημονικών μελετών να μετρήσουμε, να σταθμίσουμε, να δούμε ποιο είναι το μέγεθος, η εμβέλεια του προβλήματος και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι μικρή υπόθεση 1200 εκτάρια. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι οι αναφέροντες όπως και η έκθεση πήγαν προς την ορθή κατεύθυνση, ακολούθησαν τη σωστή πορεία. Η καλύτερη προστασία, η καλύτερη προστασία για το περιβάλλον είναι να μην αποκρύψουμε τίποτα, να αποκαλυφθούν όλα. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν που πρέπει να επιληθεί και πρέπει να επιληθεί με το συντονισμό όλων των θεσμικών οργάνων. Και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε μια ανησυχία, σε ένα μέλημα, μια ανησυχία που και η κυρία Γκρίνι το γνωρίζει πολύ καλά και είναι η σύσταση του ότι το σύνολο των μελετών που έχουν γίνει από πλευρά των επιστημονικών μελετών, επιδημολογικών μελετών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι η λιδία λίθος αυτό βρίσκεται επί Αυτό έχουμε λοιπόν από πλευράς ε, επιστημονικών μελετών. Πρέπει να εργαστούμε με βάση αυτές τις συστάσεις. Και είναι συστάσεις οι πιο σημαντικές ε, και που γίνονται αποδεκτές από τους πολίτες της Βουέλβα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ότι υπάρχει υψηλή θνησιμότητα. Είναι μια ζώνη ανώτατου κινδύνου επιδημιολογικού. Όμως δεν επεξηγούνται όλα αυτά. Για ποιους λόγους, ποια είναι τα αίτια. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες, κανένα δεν μπορεί να πει ότι έχουν ε, επιληθεί τα προβλήματα. Υπάρχει ένα επιστημονικό κενό στο οποίο πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και η κυρία Γκρίνη είναι αυτό το οποίο πολύ καλά συνοψίζει με ε, τον τρόπο που το έκανε στα συμπεράσματά της. Υπό αυτό το πρίσμα, από τη δική μου ομάδα, στα συμπεράσματα λοιπόν, στις συστάσεις για αυτή την έκθεση, βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση αυτά τα στοιχεία. Διότι το Ευρωκοινοβούλιο αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και με τις συστάσεις είναι να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος. Υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να επιληθεί. Και πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Θέλω να υπογραμμίσω και ολοκληρώνω αυτό σε σχέση με τις ε, συστάσεις, κάτι το οποίο έθεσε η κυρία Γκρίνη με πολύ σωστό τρόπο. Και αυτό είναι η ανάγκη, οι λύσεις ε, να είναι από κοινού λύσεις, ε, να επιτραπεί στους αναφέροντες η συμμετοχή, να επιτραπεί να επισκεφθούν οι αναφέροντες σε αυτή την επίσκεψη, να γίνει αυτή η επίσκεψη που δεν επετράπη στο παρελθόν με ανεξάρτητους επιστήμονες, επιστημονικό ε, προσωπικό ανεξάρτητο για να μπορέσουν να εξευρεθούν τρόποι να υπάρξει συνεισφορά για την τελική επίλυση του προβλήματος. Με τα χίλια τόσα εκτάρια να δούμε τι θα γίνει που έχουν εμολυνθεί. Για αυτούς όλους τους λόγους λοιπόν ολοκληρώνω. Κυρία Γκρίνη, συγχαρητήρια σε εσά από μένα και ελπίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, εφόσον είναι δυνατόν κάποια πράγματα να βελτιωθούν, θα προσπαθήσουμε με τροπολογίε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα. Είναι μια έκθεση που πάει στη σωστή κατεύθυνση και μα δίνει ικανοποίηση και δίνει, θα λέγα, και ικανοποίηση στου αναφέροντε. Και από κοινού με τι ε, κρατικέ αρχέ θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε να επιληθούν τα προβλήματα. Λυπούμε για το ότι δεν έχει δώσει ακόμα η Ισπανική κυβέρνηση στην ε, ε, προειδοποιητική επιστολή και εξετάζει το θέμα. Ελπίζω ότι και αυτό το ζήτημα θα επιληθεί. Εν πάση περιπτώσει το Ευρωκοινοβούλιο είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γιάννης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, η πρώτη επιτυχία αυτής της αποστολής είναι το πώς άλλαξε το κλίμα, η ατμόσφαιρα που από την επίσκεψη στην Ουέλβα μέχρι τη σημερινή συζήτηση, κυρία Γκρούνη, και εγώ προσθέτω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια που σας απευθύνθηκαν για αυτή την έκθεση και για τα συμπεράσματα και για την υπομονή και τις καλές προθέσεις που είχατε σε σχέση με την επίσκεψη στη Ουέλβα. Και λέω άλλαξε το περιβάλλον. Γιατί? Διότι εκεί υπήρχε και πρέπει να το αναγνωρίσουμε μεγάλη ένταση. Μεγάλη ένταση περιβαλλοντικών θεμάτων και μεντιατική όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και πολιτική πίεση σε σχέση με τους αναφέροντες, τους εργαζόμενους, ε, καθένας από την πλευρά του και με τις επιτροπές ε, των εργαζόμενων στις ε, βιομηχανίες αυτές και με τις επιτροπές όλα αυτά δημιούργησαν κάποια ένταση σε σχέση με την αποστολή των μελών της αντιπροσωπείας και σχεδόν θα μπορούσε κανείς να έχει χάσει, να έχανε και την ψυχραιμία του από τόση ένταση. Όμως ε, ήταν καλό α, το ότι έγινε αυτή η αποστολή. Σήμερα κάνουμε λόγο και συζητάμε υπό διαφορετικό πρίσμα, σε διαφορετικό πλαίσιο, μέσα σε ένα διαφορετικό περίγυρο και ατμόσφαιρα. Στο σημείο 3, σε σχέση με την έκθεση, αναφέρεται, η, συνοψίζεται η κατάσταση και για να αποφύγουμε καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ένα κλίμα τοπικού πανικού, έκρηξης τοπικού πανικού όσον αφορά τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να δείξουν μεγαλύτερη σύνεση στον τρόπο με τον οποίο θα επικεντρώνονται στο πρόβλημα. Μια και μια ας το πω έτσι προκλητική στάση τοποθέτηση μπορεί να είναι αρνητική όταν έρχεται η στιγμή να αναζητηθεί μια λύση αποτελεσματική και σωστή για ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό είναι που είχαμε τώρα, τώρα ε, τότε. Σήμερα όμως έχουμε προχωρήσει και έχει αλλάξει το κλίμα. Και σε σχέση με την ε, επικεφαλής του Δήμου, όπως εκφράστηκε ήταν ένα ε, μέλημα το οποίο συμμεριζόμαστε καθώς επίσης και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Γουέλβα για τη δημιουργία ενός κλίμα, κλίματος ε, πανικού που δεν θα ήταν και όλας και δικαιολογημένο και πρέπει να αποσταλεί ένα μήνυμα καθησυχαστικό ε, και με την έκθεση αυτή που έχει υποβληθεί και με τη σημερινή συζήτηση κατευθυνόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα, να κάνουμε λόγο για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικά ολέθριο, καταστρεπτικό και που επιδεινώνεται. Κάνουμε λόγο για ένα πρόβλημα το οποίο το θέτουμε στους όρους του προβλήματος που θα μπορεί να τύχει επίλυσης και που βρισκόμαστε στην τελική φάση επίλυσης. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτή την τελική φάση ώστε επαρκώς να υλοποιηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Υπενθυμίζω σε αυτή την αποστολή σε μια μικρή έκθεση που διάβασα εσωτερικά στην ειδική μας αντιπροσωπεία είδα ότι υπήρχαν δύο τύποι αντίδρασης. Ο τρόπος συναισθηματικής αντίδρασης αισθηματικά φορτισμένης και ο αντικειμενικός ορθολογικός τρόπος. Και σε σχέση λοιπόν με την αισθηματική φόρτιση σε σχέση με τους αναφέροντες και σε σχέση με την δέσμευση αυτών που είχαν επαναληφθεί στο παρελθόν όμως η ορθολογική παρέμβαση είναι εκείνη η οποία αφορά τον επιστημονικό χαρακτήρα και την επιστημονική δράση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών και στα πανεπιστήμια και στη Γουέλβα και στη Γρανάδα και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα συνεισφέρουν ώστε να μην υπάρξει σύγχυση όσον αφορά τα αίτια και και το αποτέλεσμα και το τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα από τα απόβλητα για την υγεία καρκινογένεση ή ε, προβλήματα αναπνευστικά που μπορεί να υπάρχουν στην επαρχία της Γουέλβα. Και κυρίως εμένω και επιμένω στα μέτρα που λαμβάνονται από τις κρατικές αρχές και από τις επιχειρήσεις με εντολή των κρατικών αρχών που βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση και είναι επαρκή. Νομίζω ότι έγιναν καλά τα πράγματα στην αποστολή αυτή που κάναμε και σε αυτό συμπίπτω με τον κύριο Βίλι Μάγερ. Βαίνουμε, πηγαίνουμε προς την ορθή κατεύθυνση και είναι ένα θέμα αυτό στο οποίο ευτυχώς βρισκόμαστε σε έγκαιρη αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος. Κάτι άλλο πρόεδρε και δεν ζητώ να γίνουν άλλες αποστολές. Είναι η μόνη αποστολή που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια επιχείρηση φωσφο... που παράγει ε, παράγωγα φωσφόρου. Και υπάρχει και το είδαμε αυτό στις εκθέσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις ε, παρόμοιου τύπου που παράγουν ε, λι... λιπάσματα σε άλλες έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, καμία δεν ελέγχθηκε ή δεν επιθεωρήθηκε ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από την Ευρωβουλή. Καμία δεν υλοποιεί από αυτές ε, τις ε, διατάξεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση και ανάλυση όπως γίνεται από αυτές τις επιχειρήσεις ε, της Μπάτσαντε Φασαουέφος της Γουέλβα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι με βάση αυτό αυτή την πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια στην ε, Γουέλβα, αυτή η τεχνολογία που υιοθετήθηκε είναι μια τεχνολογία που μπορούμε να συστήσουμε να εξαχθεί σε άλλες ε, επιχειρήσεις λιπασμάτων, παραγωγής λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο πρέπει να γίνει είναι να εφαρμόσουν τους μηχανισμούς ελέγχου όπως γίνεται από τη Γουέλβα Αυτά είναι τα συμπεράσματα του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Όκεν. Εγώ θα είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Πασκάλα Γκρουνή για την έκθεση που μας έκανε. Εντάξει, μπορώ να την ευχαριστήσω μετά. Ακούγοντας τις διάφορες ε, παρεμβάσεις, ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι ότου να καταφέρουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι εκεί με έναν ευγενή ε, και πολιτισμένο τρόπο ώστε να μπορέσουν δηλαδή να συνομιλήσουν. Πρέπει να πούμε για τη βελτίωση της επικοινωνίας γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση εδώ ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη. Είμαι ικανοποιημένη λοιπόν από την έκθεση και ικανοποιημένη από τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Αποδείξαμε ότι, χρειαζο... ότι μας χρειάζονται φέτος, λοιπόν. Grazie. Σας ευχαριστώ. Eh, Θέλω να απαντήσει η κυρία Πέτρο Γκερέρο Ροζάντο. Να της δώσω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να παρέμβω. για να προσπαθήσω κατά κάποιο τρόπο να απαντήσω σε ορισμένα από τα πράγματα που αναφέρθηκαν εδώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μέγερ ότι δεν πρόκειται για καμία προσπάθεια ε, συγκάλυψης. Αντίθετα, ε, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την πόρτα στην επαρχία της Ουέλβα, στην κυρία Γκρούνη και στην Κομισιόν Νομίζω πως ε, κάτι τέτοιο δικαιώνει την πραγματικότητα που ισχύει στην ε, περιοχή μας. Υπάρχει ένα θέμα. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Ο εκπρόσωπος ε, της Μέσα Ντελαρία μίλησε στο παρελθόν, στον αόριστο και περιέγραψε μια πραγματικότητα 20-25 ετών. Όπως σας είπα και στη δική μου παρέμβαση, όταν ήρθατε στην Ουέλβα και ακόμα και σήμερα ζήτησα συγγνώμη στην κυρία Γκρούνη για το συμβάν που έγινε γιατί για δεύτερη φορά δεν μπορέσατε να επισκεφτείτε το χώρο απλούστατα γιατί δεν είχατε ζητήσει την έγκριση από την επιχείρηση, από το εργοστάσιο. Και φαίνεται ότι θα ήταν ανεύθυνο να επιτραπεί η είσοδος ενός ατόμου που δεν ε, είχε την απαραίτητη άδεια. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ποια είναι η κατεύθυνση που έχουμε ακολουθήσει για την επαρχία της Ουέλβα. Η αρχή ορυπαίνων πληρών προβλέπεται για αυτού του είδους τα προβλήματα. Η επιχείρηση θα πρέπει να βρει μια λύση στα θέματα στα προβλήματα ρήπανσης. Ε, σε ένα μήνα θα γνωρίζουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ε, πιλωτικής έρευνας που έγινε, γιατί ο χώρος αυτός αποτελεί ε, πλέον ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα, γιατί επιτρέπει να δημιουργηθούν και παραπάνω θέσεις εργασίας. Και πάλι κυρία Γκρούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την δουλειά σας. Η έκθεσή σας δικαιώνει την πραγματικότητα που ισχύει στην επιαρχία της Βουέλβα. Κάνετε μια σειρά από συστάσεις με τις οποίες ε, συμφωνώ, ιδιαίτερα εκείνη που συστήνει να μην δημιουργηθεί πανικός, να μην ε, δυναμητιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να φτάσουμε σε μια οριστική λύση. Τέλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν γίνεται ή όχι, αλλά θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους να έρθετε, να δείτε την, να γνωρίσετε την επαρχία μου. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να σας υποδεχτώ εκεί, ώστε να μπορέσετε να εκτιμήσετε τον αριθμό των ηλιόλουστων των ημερών που έχουμε και τις ε, παραλίες, τις υπέροχες παραλίες που έχουμε στην ε, επαρχία μου. Σας ευχαριστώ και ε, ελπίζω να σας δω σύντομα στην Ουέλβα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Πέντρου Χιμένε ζήτησε το λόγο. Έχω τρία πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο Φαντάζομαι ότι όταν η κυρία της αντιπροσωπείας μιλά, είμαστε δύο εκπρόσωποι της Μέσα Ντελαρία. Μία, ένας από την ε, σύνδεσμο και άλλος ε, από την πλατφόρμα και οι δύο είμαστε αναφέροντες. Φαντάζομαι ότι αναφερθήκατε σε μένα γιατί παρατηρήσατε ότι όσα έχετε γράψει είναι πραγματικότητα σήμερα και μπορέσετε να διαπιστώσετε παρά τα εμπόδια που συναντήσατε ως αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Ουέλβα. Εκεί που σας απαγορεύθηκε η είσοδος είναι δημόσια ε, χερσαία και θαλάσσια περιοχή που αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί από μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι δηλαδή χώρος όλων, έδαφος όλων, δημόσιο έδαφος. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό να το διευκρινίσουμε. Και το να, να λένε ότι οι αναφέροντες δεν ζήτησαν έγκριση για να επισκεφθούν τη Φερτιμπέρια είναι επειδή στην Ουέλβα κανονικά μπορούσαμε να επισκεφτούμε οποιοδήποτε μέρος τέτοιο χωρίς πρόβλημα. Δεν υπάρχει ούτε λουκέτο, ούτε κανένας ε, φύλακας που να μην επιτρέπει να μπούμε εκεί. Και επιπλέον, ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν την συγκεκριμένη τοποθεσία και θα έπρεπε να μπορούν να μεταβούν εκεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εγώ έχω φωτογραφίες παλιότερες, μπορώ να σας δώσω την ακριβή ημερομηνία όπου έγινε αυτό. Στόχος είναι μόνο η ίδια η εταιρεία να εμποδίσει την επίσκεψη από πλευρά των Ευρωβουλευτών. Μια πολύ απλή ερώτηση τώρα για δύο πράγματα. Καθώς σήμερα όλοι είναι πολύ ικανοποιημένοι και ολοκληρώνω από την επίσκεψη που έγινε στην Ουέλβα θα μπορούσα ωστόσο να σας στείλω πολλά αποσπάσματα του τύπου όπου πολλοί πολιτικοί ηθήνοντες της ε, ΟΕΛΒΑ αλλά και συνδικαλιστές κατηγόρησαν τους αναφέροντες για το ότι η Επιτροπή Αναφορών επισκέφθηκε την Όλβα, ότι δηλαδή εμείς ε, αμαυρώσαμε την εικόνα της ΟΕΛΒΑ. Είναι μια πραγματικότητα που, δυστυχώς, ε, που ευτυχώς σήμερα έχει ξεπεραστεί. Καμιά μελέτη και ολοκληρώνω και ζητώ και συγγνώμη, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει το τη σχέση αίτιου και αιτιατού για τις, ε, τους θανάτους από το καρκίνο. Υπάρχουν όμως ε, μελέτες, ούτε και υπάρχουν μελέτες που ε, να αποδεικνύουν το αντίθετο. Δηλαδή καμιά μελέτη που δεν έχει γίνει που έχει γίνει εκεί από τον καθηγητή Βενάν και το Πανεπιστήμιο της περιοχής όπου λέει ότι ο δείκτης καρκίνου καρκινογένεσης είναι 15% ψηλότερος από οπουδήποτε αλλού. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε κύριε. Ο κύριος Ντάβιτ Χάμερστεν. Εγώ ήθελα να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον και είμαι ευτυχής που μιλήσαμε για το μέλλον και για έναν πράσινο πνεύμονα της πόλης αλλά όταν μιλάμε για απορρίπανση, δεν μπορούμε να πάρουμε τα ίδια μέτρα όπως η BP με το ατύχημα στο κόλπο του Μεξικού και να στείλουμε άλλες χημικές ουσίες για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και να σταματήσουμε την διαρροή. Δεν μπορούμε να καμουφλάρουμε την κατάσταση φυτεύοντας κάποια φυτά εκεί, κάποια δέντρα και ελπίζοντας ότι θα ενεργήσουν ως απορριπαντικοί παράγοντας. Όχι. Καταρχήν <coughs> θα πρέπει να ακολουθήσουμε υποδειγματικούς τρόπους να ε, ε, κατεργαστούμε και να μεταφέρουμε τόνους τοξικών αποβλήτων θα επιτρέψει να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα είναι ένα παραπάνω πλεονέκτημα για την απορρίπωση. και αυτό που εγώ προσωπικά ζητώ από την Επιτροπή Αναφορών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις αρχές της Βουέλβα είναι να ζητήσουν μια αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να απορριπάνουμε την περιοχή και να ζητήσουμε για παράδειγμα μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη για το πώς θα μπορούσε να καθαριστεί εις βάθος η περιοχή και όχι μόνο επιφανειακά. Έπειτα, σε σχέση με την έκθεση αιτίου αιτιατού για την ύπαρξη αυτών των ουσιών και τις καρκινογενέσεις. Δεν υπάρχει μόνο ένα αίτιο, για παράδειγμα, καρκίνο. Υπάρχουν πολύ περίπλοκες διαδικασίες και μείγματα ουσιών που μέσα σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο έχουν επιπτώσει στην υγεία ατόμων και προκαλούνται έτσι αλλού περισσότερες περιπτώσεις, αλλού λιγότερες ε, καρκινογενέσεων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αντικειμενικοί και να γίνουν αυτές οι μελέτες από ανεξάρτητους επιστήμονες που δεν θα έχουν καμιά σχέση με βιομηχανίες ούτε με άτομα που είχαν επαφή με κάποια άλλα. Αυτό λοιπόν αυτό το οποίο ζητάμε είναι να αντιμετωπιστούν τα απόβλητα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πανικό. Θέλουμε να μπορούμε να αγαπάμε τις, ε, τη γη και τα άτομα άτομα και να τα προστατεύουμε. Να μην υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα... δεν είναι τα άτομα που μολύνουν ε, την περιοχή της Βουέλβα. Είναι τα απόβλητα τα οποία μολύνουν εδώ και δεκαετίες στην Βουέλβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφος Γιάννης. Συγγνώμη πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο μόνο και όχι για όλα τα θέματα αλλά για το συγκεκριμένο εξειδικευμένο το οποίο αναφέρθηκε στο τέλος και στο οποίο είχα αναφερθεί όσον αφορά το θέμα του αίτιου και του αιτιατού. Και πέρα από ευρωβουλευτής, πέρα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είμαι γιατρός. Ξέρω διπλά για τι πράγμα κάνω λόγο. Εδώ σε περιπτώσεις καρκίνου που είναι ε, επίκαιρη υπόθεση ο καπνός έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι αίτιο του καρκίνου των πνευμόνων. Δεν είναι κάτι το οποίο αποδείχθηκε ε, σήμερα είναι κάτι το οποίο το 1968 αποδείχθηκε από Βρετανούς επιστήμονες. Στο παρελθόν πριν από αυτήν την ημερομηνία υπήρχαν υποψίες, αλλά χωρίς καμιά αμφιβολία από τα τέλη της δεκαετίας του 60 έχει αποδειχθεί. Είναι ένας συσχετισμός αιτίου και αιτιατού. Ο καπνός, το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Και εδώ σε σχέση με το αν υπάρχει κάποιο συσχετισμός αίτιου αιτιατού για τις περιπτώσεις καρκίνου στη Γουέλβα δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία τώρα μπορεί να υπάρξει κάτι στο μέλλον. Εγώ αναφέρθηκα στο πώ έχει η πραγματικότητα σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, Και εγώ θα ήθελα να κάνω λόγο για αυτό το θέμα, διότι είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα αναφέρεται. Αναφέρεται από πλευρά των ε, επιστημόνων, αναφέρονται στοιχεία, αναφέρονται άλλα στοιχεία από την Γουέλβα. Τα επιδημιολογικά, επιστημολογικά στοιχεία. Είμαστε πολύ πάνω από το μεσόωρο. Η επιστημονική ε, κοινότητα δεν μπορεί ακόμα να το πει. Γιατί συμβαίνει αυτό. Οι πολίτες διεκδικούν και θέλουν εξηγήσει και ζητούν να υπάρξει επίρρηψη ευθυνών. Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να γίνεται είναι να μην αποκρύβονται στοιχεία. Με την αποκάλυψη στοιχείων πρέπει να αποκαλυφθεί το τι συμβαίνει. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα πολύ περίπλοκο. Δεν είναι στατιστικά στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε να επαρκέσουμε πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο κάθε μια από τις περιπτώσει αυτέ, Είναι ένα πολύ μεγάλο περίπλοκο θέμα. Και υπάρχει και σε σχέση με το, ε, την, την περιοχή και του Γιβραλτάρ και από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητηθεί από τις Ισπανικές αρχές και από τις Βρετανικές αρχές να υπάρξει μια επιδημιολογική επιστημονική μελέτη σε αυτή τη ζώνη ώστε η απουσία αυτών των βεβαιοτήτων να αντιμετωπιστεί με επιστημονικά αντικειμενικά στοιχεία το α, το β, το γ να δράσουμε έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα αποσαφήνισης και διευκρίνησης περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρούνη θέλει να παρέμβει παρακαλώ. Ναι. Δύο λόγια. Γιατί έκαναν λόγο για την επίσκεψη που δεν έγινε με τους αναφέροντες ε, επιτόπου στον χώρο του εργοστασίου. Είναι ένα θέμα, όπως σας είπα, εξαιρετικά λεπτό και προσπάθησα να ηγηθώ της αντιπροσωπείας ε, με μεγάλη νυφαλιότητα, πράγμα το οποίο δεν ήταν πάντοτε προφανές, όπως θύμισε ο κύριος Γιάννης. Και όταν φτάσαμε εκεί με τους αναφέροντες, ε, είχε ένα σωρό κάμερες εγώ αρνήθηκα λοιπόν να προχωρήσω γιατί εκεί θα γινόταν μια επίσκεψη που θα ήταν τελείως διαφορετική. Ε, ωστόσο πιστεύω πως η επιχείρηση έχει κάθε συμφέρον να ε, ενεργήσει με διαφανή τρόπο, να επιτρέψει να γίνει η επίσκεψη με τους αναφέροντες και εκπροσώπους για να πάνε να δουν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα σημεία που είναι προβληματικό το θέμα για τους αναφέροντες. Είναι αλήθεια για τις μελέτες είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι καταρχήν όταν γίνεται λόγος για καρκίνο και ο κύριος Γιάννης το θύμισε επίσης, Εμάς μας είπαν σε επιτόπου ότι αυτή η περιοχή είχε ένα ποσοστό ραδιενέργειας πιο υψηλό από ό,τι αλλού και ότι θα μπορούσε ε, αυτό να ισχύει και πριν να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα ή συμβάν. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι δύσκολο το θέμα. Οι μελέτε θα πρέπει να γίνουν, πιστεύω, με τρόπο συντονισμένο, με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, για να υπάρχει εμπιστοσύνη στις μελέτες αυτές. Σήμερα ο κ. Γενές μίλησε για τον καρκίνο του πνεύμονα. Γίνεται λόγος επίσης για τον παθητικό καπνιστή και πριν από δύο μέρες μας είπαν ότι ο παθητικός καπνιστής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ενώ εδώ και πολλά χρόνια μας λένε ότι ο παθητικός καπνιστής μπορεί να, έχει τον ίδιο καρκίνο, να πάθει τον ίδιο καρκίνο όπως αν κάπνιζε. Οπότε δεν υπάρχουν βεβαιότητες, ωστόσο υπάρχει και επικοινωνία και εδώ στρέφουμε και στην, προ... στην ε, τις περιφέρειες που είναι σήμερα μόνη της εδώ, αλλά φυσικά αυτό ε, το, απευθ... το αίτημα το, ευθύνω... απευθύνω σε όλους ε, τους ηθήνοντες στην Ισπανική Αρχή. Ε, συστήνω διαφάνεια, απορρίπανση του χώρου, να εξεταστεί η δυνατότητα απορρίπανσης, να τεθεί φυσικά και η επιχείρηση ενώπιον των ευθυνών και εγώ σα λέω ευνίδιοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται. Σα διαβεβαιώ πω αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και τέλο, ε, ε, καταλάβαμε και αισθανθήκαμε πως υπάρχει ανησυχία από πλευράς του πληθυσμού και γι' αυτό και ακριβώς ε, υπήρξαν πολλές αναφορές ε, που ακόμη και σήμερα ε, υποβάλλονται, αλλά εμείς ήρθαμε σε επαφή και με ανήσυχους υπαλλήλου, υφευθύνου των συνδικάτων που ανησυχούν για, την, ε, για τη δουλειά τους και θα πρέπει να, κανείς να ακούσει όλους και να βρει την καλύτερη λύση και φυσικά θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Γκρούνη για την εξαιρετική σας εργασία. Ευχαριστούμε για τους αναφέροντες, τους που παρενέβησαν και θα αναβάλουμε οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα έχουμε το χρόνο για να το σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε την